Let's start, even if there a problem, there is a problem. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει ε, πρόβλημα για πολλούς συναδέλφους ε, να έρθουν στις Βρυξέλλες. Ε, και εγώ είχα πρόβλημα. Ήθελα κανονικά να έρθω από χτες το βράδυ, τελικά τα κατάφερα να έρθω, να έρθω σήμερα στις 3. Πάλι καλά, γιατί έχουμε πολλές καταιγίδε. Πάμε λοιπόν στην έγκριση της σημερινής διάταξης έχουμε το 4, θα συζητηθεί μετά το 15, ε, το οποίο 15 ε, το έχετε μπροστά σας, θέσπιση του μηχανισμού προνταξιακής βοηθείας. Αν δεν, ε, δεν διαφωνείτε, τότε εγκρίνεται αυτή η πρόταση που κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο εξή. Η απόφαση των συντονιστών της 13 Σεπτεμβρίου βρίσκονται ήδη τα πρακτικά ε, καταχωρημένα, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται και αυτά. Και πάμε στην έγκριση των πρακτικών της 26ης Ιουνίου του 2018. Δεν ξέρω αν έχετε αντιρρήσεις, από ό,τι βλέπω όχι. Ως εκ τούτου εγκρίνεται και αυτό το θέμα. Και μπορούμε να περάσουμε στην ε, σύσταση του προγράμματος για την ε, θέσπιση του προγράμματος Τελωνία για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνίων. Ο Στάλφος Στέφανεκ, από ό,τι βλέπω, έχει φτάσει. Ε, πολύ καλό αυτό και έτσι διευκολύνει και η κατάσταση. Έχετε το λόγο. Ε, μιλάμε για το να υπάρχει ένα πρόγραμμα τελωνιακό στον τομέα των τελωνίων. Και κατ' ουσίαν μιλάμε για τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήματα υπολογιστών στα κράτη-μέλη και το να συσταθεί το πρόγραμμα αυτό μετά το 2020, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να προστατευτούν ε, τα συμφέροντα των τελωνίων και των κρατών μελών. Έχουμε 950 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2021 ε, και αυτό να ελοπιθεί το πρόγραμμα μέχρι το 2027. Αυτό είναι το ποσό. Κατ' ουσίαν προβλέπεται να ε, εγκατασταθούν συστήματα, συμβατά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα τελωνία καλούνται να εξετάσουν το κατά πόσον αυτά θα είναι αρμονικά με άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόγραμμα Φισκάλης, το πρόγραμμα για την, κοινή αγορά, το πρόγραμμα για την ψυχιακή Ευρώπη, Connecting Europe Facility και αποφάσει σχετικά με τους ίδιου πόρου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μια πολύ καλή βάση και εγώ στηρίζω την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί, λέει πρόεδρο, Άιντα, εσείς είστε σκαιώδης εισηγήτρια, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δύο φράσεις μονάχα γιατί υποστηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν και συμφωνούμε και με τα όσα αναφέρει ο εισηγητής. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Is there anybody... Κανείς άλλος επιθυμεί, κάποιος άλλος ενδεχομένως να πει κάτι ως σκιώδης εισηγητής με αυτή του την ιδιότητα. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια από άλλες ομάδες ε, κατόπιν τούτου. Θα ήθελα να σου θέλετε να προσθέσετε κάτι. Από ό,τι βλέπω όχι. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 3η Οκτωβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμών θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου Βλέπω συμφωνείτε και δεν βλέπω να έχουν έρθει οι συναδελφοί μου για τις επόμενες δύο γνωμοδοτήσεις. Ως εκ τούτου θα ήθελα να περάσουμε στα θέματα της κτηριακής πολιτικής και ίσως ε, με τον τρόπο αυτό μπορούμε και να καλύψουμε το κενό που υπάρχει τώρα στην Επιτροπή. Θα μιλήσω γερμανικά βέβαια. Αλλά μιλάω αγγλικά mm το κοινοβούλιο ε, αγόρασε το σπίτι Ζαν Μονέ στο Μπαζός ε, το 2018. Ε, Εδώ λοιπόν στην Επιτροπή Προπολογισμών ήδη συζητήσαμε, έχουμε συζητήσει για το κτίριο αυτό και τότε είχαμε ήδη καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, το κτίριο αυτό να το χρησιμοποιεί περισσότερο για συνέδρια και παρεμφερείς εκδηλώσεις. Ε, κάτι το οποίο όμως ήταν αρκετά δύσκολο διότι υπήρχαν προβλήματα φιλοξενίας. Το 2018 λοιπόν αγοράστηκε το κτίριο αυτό, το 2012 ανακαινίστηκε, το 2016 ε, ολοκληρώθηκε το συνεδριακό κέντρο και υπάρχει η ανακοίνωση ενός γείτονα το 2017 για την πώληση του γειτονικού οικοπαίδου και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας αν θέλαμε να χρησιμοποιούμε το συνεδριακό κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έπρεπε λοιπόν να αγοράσουμε και αυτό το γειτονικό οικόπεδο. 1.200 ε, τετραγωνικά μέτρα, 60.000 ευρώ το σύνολο, άρα ε, το ποσό είναι αρκετά ικανοποιητικό και η τιμή κυμαίνεται από 108 μέχρι 234 ευρώ, άρα είναι ικανοποιητική η τιμή. Βέβαια, έχουμε κάποια έξοδα συμβολογράφου, τα οποία αυτή τη στιγμή τα βρίσκω αρκετά υψηλά, εγώ τουλάχιστον. Ε, νομίζω ο συνάδελφος Dupré, ε, ρώτησε και ήθελε να μάθει ε, ποια θα είναι ακριβώς η χρήση αυτού του κτηρίου. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ που να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο και να μπορεί να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Από ό,τι βλέπω το Κοινοβούλιο ε, αυτή τη στιγμή έχει διάλειμμα, ίσως έρθουν αργότερα. Αν συμφωνείτε και εσείς να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Κατόπιν πάμε στην εκμίστοση του κτηρίου Eurooffice στο Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή το κτίριο, μέχρι να γίνει η μετακόμιση στο νέο κτίριο, πρόκειται για συμπληρωματική εκμίστοση μέχρι την ολοκλήρωση του νέου κτηρίου επέκταση του μισθωτηρίου συμβολέου το Λουξεμβούργο, το κράτος του Λουξεμβούργο είναι, ε, συνυπογράφει το συμβόλαιο αυτό. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία αύξηση του μισθώματος που το βρίσκω παράδεικτο. Γιατί το να ζητάει κανείς αύξηση της τάξης του 46% είναι ανέδεια. Και πρέπει να το επισημάνουμε ότι ε, εμείς παλαιότερα είχαμε καταβάλει ένα ποσό που ήταν βέβαια πολύ χαμηλό. Με πάση περιπτώσει ε, αυτή την ε, τερατώδη αύξηση τη βρίσκω όπως σας είπα γένεια. Από ό,τι φαίνεται υπήρξαν κάποια προβλήματα στις ε, διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να ρωτήσω το Κοινοβούλιο, αυτό το 46% πώς το εξηγείτε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια καλύτερη προσφορά έστω και αν αυτό που πληρώναμε παλαιότερα πράγματι ήταν κάτω από το ε, μίστομα το οποίο θα έπρεπε να έχουμε καταβάλει. Μία ερώτηση προς την ΟΕΛ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου θέλουμε ε, να παραμείνουμε για κάποιο διάστημα ε, στο κτίριο Eurofis ε, Mercier για τέσσερα χρόνια. Αυτό θα μας επιτρέψει αργότερα να έχουμε τη δυνατότητα να νοικιάσουμε και να, να έχουμε τα γραφεία μας στο Mercier Post. Ε, το προηγούμενο κτίριο πρόκειται να ε, ε, να κατεδαφιστεί. Ε, και επομένως, όντως το ενίκιο ε, είναι 18 ε, ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα. Ήταν η αρχική συμφωνία πριν από πάρα πολλά χρόνια στο αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο και οπωσδήποτε είναι εκτός αγοράς αυτή τη στιγμή. το είπατε και εσείς αυτό και αυτό εξηγεί και την μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο παλαιό ενίκιο μίσθωμα και στο νέο και το νέο μίσθωμα εξακολουθεί να είναι κάτω από τις ε, τιμές αγοράς του Λουξεμβούργου. Η διαφορά κατ' είναι 2,7 εκατομμύρια, για να το πω έτσι απλά και καθαρά. Ναι, έχετε απολύτως δίκιο, αλλά πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το παλαιό κτίριο. Χρησιμοποιούμε ε, λιγότερη επιφάνεια, ε, περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ε, και θα, φτάσουμε, θα κατεβούμε στα 23 ανά κάτοχο και επομένως είναι και ένα ποσοστό εκμετάλλευσης χαμηλότερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Ε, εσεί εσείς στο νέο κτίριο, το οποίο θα κοστίσει 9,37 εκατομμύρια. Τώρα στα 10, κάτι. Ε, άρα δηλαδή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με αυτό το ε, συμπληρωματικό ε, συμβόλαιο θα έχουμε μια ουσιαστική αύξηση από τα 9 τόσα θα πάμε στα 10 τόσα εκατομμύρια νομίζω ότι αυτό ε, δεν είναι τόσο ευνοϊκό όσο θα έπρεπε να υπάρχει με το συμπληρωματικό σύμβολο. Και θέλω να ρωτήσω, εφόσον είναι έτσι κι αλλιώ ένα παλιό κτίριο, δεν υπάρχει δυνατότητα κάπως να ασκήσουμε πίεση στον ε, εκμισθωτή, γιατί ζητάει μια αύξηση της τάξης των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σας λέω, τερατώδης αυτή η αύξηση. Ένα κτίριο το οποίο θα έχουμε με συμπληρωματικό συμβόλαιο. Και με τα ενοικίαση του άλλου κτιρίου, το Monsieur Post, εκεί η συνολική έκταση θα είναι μικρότερη, θα είναι 16.077 τετραγωνικά μέτρα. Ε, πιο, αποτελεσματική, πιο αποτελεσματικό θα είναι αυτό το κτίριο. Ετήσιο ε, κόστος 6,9 εκατομμύρια ευρώ, 424 ήταν περίπου ε, ανατετραγωνικό. Ε, είναι λιγάκι ακριβό, πρέπει να σας το πω αυτό αγαπητοί Κομισιόν, κάπως να τα βρείτε λιγάκι με το κράτος του Λουξεμβουργού, γιατί αυτή είναι πολύ πιο ακριβή από ό,τι εδώ στις Βρυξέλλες, μα πάρα πολύ πιο ακριβή. Όταν λοιπόν θα κληθούμε να συγκρίνουμε το συνολικό κόστος στο συμπληρωματικό ε, συμβόλαιο θα έχουμε 10 κόμμα τόσα συμπεριλαμβανομένων ε, και τα πάγια, ε, τις πάγιες δαπάνες. Αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αποδεκτό. Εσείς δεν βλέπετε να υπάρχει καμία δυνατότητα στο συμπληρωματικό μισθωτήριο συμβόλαιο να πείσουμε τον εκμισθωτή ε, να μας ε, δώσει μια καλύτερη, ε, μια καλύτερη πρόταση, γιατί σας είπα, το 46% είναι για μένα απαράδεκτο μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί κατά το παρελθόν πληρώναμε συμβόλαιο, είχαμε συμβόλαιο και πληρώναμε μισθώμα κάτω του κόστους. Απάντηση. Όσον αφορά ε, την ε, χαμηλή τιμή ε, που πληρώναμε στο παλιό κτίριο για κάποια χρόνια πρόκειται για μια τιμή η οποία συμφωνήθηκε στην υπογραφή του πρώτου μισθωτηρίου συμβολέου πριν από 30, ίσως και 40 χρόνια. Ήταν τελείως διαφορετικές οι τιμές. Ε, το κτίριο τώρα βρίσκεται στο τέλος της ζωής του. Μπορούμε, μπορεί να λειτουργήσει για μερικά χρόνια ακόμα ε, χωρίς δυσκολία. Ωστόσο, αυτή η μετάβαση δημιουργεί πρόβλημα στο business plan του ιδιοκτήτου, διότι αυτό το κτίριο βρίσκεται σε, ένα, σε μια γειτονιά ε, στην οποία θα κατεδαφιστούν και θα χτιστούν εκ νέου όλα τα παλιά κτίρια, μεγάλα κτίρια γραφείων και επομένω, καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο αυτό εμεί του δημιουργούμε πρόβλημα ε, στον σχεδιασμό του. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησε να βρούμε μια συμφωνία με μια ενδιάμεση τιμή ανάμεσα στην τιμή αγορά και την τιμή που μας ε, προτείνει. Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο, άρα και μεταβατική λύση, διότι εμεί σε λίγο θα πάμε στο Μερσιέ Πόστ, που είναι ένα ε, κτίριο δύο-τριών χρόνων, πάρα πολύ νέο, και όπου εμείς θα εγκατασταθούμε χωρίς να αναγκαστούμε να κάνουμε καμία τροποποίηση και όπου βεβαίως η τιμή είναι η νέα τιμή της αγοράς. Μεταβατική τιμή λοιπόν για μεταβατική περίοδο και στην ουσία αντιπροσωπεύει και την αποζημίωση κατά κάποιο τρόπο την οποία ζήτησε και με την οποία συμφωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη έτσι ώστε και αυτό να αποζημιωθεί ε, για την αλλαγή των σχεδίων του και την καθυστέρηση των σχεδίων του για 3-4 χρόνια. Ευχαριστώ. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι το συμπληρωματικό μισθωτήριο συμβόλαιο και το δεύτερο τμήμα είναι η εκμίσθωση του νέου κτηρίου του Μεσχεπόστα. Συμφωνείτε από αυτού παρακαλώ. Από ό,τι βλέπω συμφωνείτε όλοι. Ως εκ τούτου ας ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν επιφυλάξεις κατά του συμπληρωματικού μισθωτηρίου ε, συμβολέου. Από ό,τι βλέπω όχι. Βέβαια δεν έχουμε και πολλέ άλλε εναλλακτικέ λύσει, γιατί το να βγούμε από αυτό το κτίριο και να πάμε σε ένα άλλο κτίριο αυτό θα σήμαινε περισσότερε δαπάνε. Άρα δηλαδή είναι κανεί αναγκασμένο να συμφωνήσει ε, βέβαια με την παρατήρηση ότι αυτό το 46% είναι απαράδεκτο και στο μέλλον θα πρέπει η ΟΕΛ να κάνει καλύτερε διαπραγματεύσει. Σα το λέω ξεκάθαρα και θα το γράψω και στα πρακτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε προβλήματα με εσά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγεται. Παρακαλώ, ψηφίζουμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Α, όχι, δεν ψηφίσουμε τώρα, θα ψηφίσουμε αύριο. Πάμε λοιπόν πίσω. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου εδώ. Α, είναι από την άλλη πλευρά η εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου. Μπερδεύτηκα, λέει η Πρόεδρος. Είχα δύο ερωτήσεις σχετικά με το Monnet House. Η μία ερώτηση αφορά, προέρχεται από τον συνάδελφο ε, Ντεπρέ που θέλει να ρωτήσει το συνεδριακό κέντρο ποιος θα το χρησιμοποιεί. Και το δεύτερο ερώτημα είναι το κόστος, ε, οι συμβολογραφικές δαπάνες, γιατί αποτελούν το 1 πέμπτο του συνόλου κόστους ε, για το νέο μισθωτήριο συμβόλαιο. Λοιπόν, το κτίριο Μπαζός ε, χρησιμοποιείται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα η υποδοχή ε, των ε, επισκεπτών του οίκου Ζαμονέ. Περίπου 10.000 επισκέπτες το έτος. Επίσης, ε, υπάρχει όλος ο εξοπλισμός ο συνεδριακός έτσι ώστε να μπορούν εκεί να οργανώνονται πολλές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίως δε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ε, για τους νέους διοικητικούς ε, υπαλλήλου, οι οποίοι όλοι τον πρώτο, τους πρώτους μήνες πριν αρχίσουν την εργασία τους στο Κοινοβούλιο περνούν από μια τριμερή, τριήμερη κατάρτιση η οποία λαμβάνει χώρα στο κτίριο Επίση, Επίσης, εκεί μπορούν να συνεδριάσουν ε, κάποια καταδιαστήματα, διαστήματα, προεδρείο, ε, κάποιες γενικές διευθύνσεις κλπ. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε περίπου δύο ή τρεις ημέρες ε, χρήση του κτηρίου αναμήνα, δηλαδή περίπου 40 ημέρες ε, το χρόνο. Τις άλλες, τις υπόλοιπες ημέρες, ε, ο συνεδριακός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τις ομάδες επισκεπτών, ε, τους οποίους υποδεχόμαστε σε αυτήν την αίθουσα πριν ξεκινήσουν την επίσκεψή τους του οίκου Ζωμονέ και πριν λάβουν κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τον Ζωμονέ και το έργο του. Αυτή είναι η χρήση λοιπόν ε, του Μπαζός και του Συνεδριακού Κέντρου, της αίθουσας δηλαδή. Να σας πω ότι πριν από μερικούς μήνες ε, αποφασίστηκε ε, να εγκατασταθεί και ε, εξοπλισμός Europe Experience σε αυτόν τον ε, χώρο. Όσον αφορά τώρα τα συμβολιογραφικά, το συμβολιογραφικό κόστος, ναι, να σας πω ότι αυτά είναι τα νόμιμα ποσοστά τα οποία εφαρμόζονται και ισχύουν στη Γαλλία. Επίσης, συχνά υπάρχουν και, και τα το κόστος ε, καταχώρησης. Αυτό το κόστος καταχώρησης ε, εμείς θα προσπαθήσουμε σαν κοινοβούλιο να το αφαιρέσουμε έτσι ώστε να μείνει μονάχα η αμοιβή του συμβολιογράφου και όχι επομένως ο φόρος τον οποίον δεν καλείται ε, το κοινοβούλιο κανονικά να πληρώσει. Εκπίπτει δηλαδή κανονικά αυτός ο φόρος καταχώρησης. Ευχαριστώ. Στην 40.000 bei einem Gesamtpreis von 260.000 Euro. Euh, Απάντησή σας λέγω ε, ένα τμήμα των 40.000 ε, ευρώ θα ε, εκπέσουν και επομένως θα επιστραφούν καθότι αποτελούν το τμήμα του φόρου καταχώρησης. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν πίσω στη... Πάμε πίσω στην ημερήσια διάταξη, στις γνωμοδοτήσεις. Έχει έρθει ο συνάδελφος Μούρεζαν. Ε, σας το είπα και πριν ότι όλοι είχαμε προβλήματα να φτάσουμε εδώ. Ε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Μούρεζαν, θα ήθελα να σου δώσω το λόγο. Καλημέρα. Αυτή είναι λοιπόν η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας και η γνωμοδότηση που σας παρουσιάζω βασίζεται σε κάποιες αρχές που έχουμε συμφωνήσει από κοινού με τους συντελεστέ μας. Πρώτα απ' όλα εστιάζουμε σε θέματα προεπολογισμού. επομένως το φάσμα του Ταμείου Συνοχής είναι κάτι το οποίο θα συναποφιστεί με άλλες επιτροπές. Η δική μας η Επιτροπή εστιάζει σε ζητήματα προπολογισμού. Δευτερευόντω, ξεκινήσαμε από το ψήφισμα που εγκρίναμε από κοινού τον Μάρτιο και η γνωμοδότηση αυτή εδώ είναι η ερμηνεία σε θέματα προϋπολογισμού των όσων αποφασίστηκαν για το πολιετές δημοσιονομικό πλάνο τον Μάρτιο. Αυτό εδώ λοιπόν έχουμε μεταφράσει σε νούμερα στην γνωμοδότηση αυτή. Για να ξεκαθαρίσω Επίσης, χρησιμοποιούμε τρέχουσες τιμέ. Το ντοσιέ στο σύνολό του θέλει να αυξήσουμε από 330 δισεκατομμύρια σε 372 δισεκατομμύρια. Το ποσό επίσης προτείνω να, να διατηρήσουμε το επίπεδο συγχρηματοδότησης, άρα απορρίπτουμε ε, κατά συνέπεια την πρόταση της Επιτροπής. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποφασίσαμε από κοινού με συναδέλφους από την Ρέτζη Επιτροπή σε ό,τι αφορά την συγχρηματοδότηση. Μια άλλη πρόταση που περιλαμβάνεται στην γνωμοδότηση είναι να αυξήσουμε σταδιακά την προχρηματοδότηση από 0,5% σε 2%. Ε, Ιδίω προς τα τελευταία χρόνια του MFF, του πολιετούς δημοσιονομικού σχεδίου πλαισίου. Επίσης, προτείνω να αυξήσουμε τα επιδόματα για την ε, γεωγραφική συνεργασία από 2,5% σε 3%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία. Ένα άλλο στοιχείο που περιλαμβάνεται στη γνωμοδότησή μου είναι κάτι το οποίο ως κοινοβούλιο ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια. Τα ποσά δηλαδή δεν πηγαίνουν απευθείας στα κράτη-μέλη, αλλά παραμένουν σε ένα κοινό ταμείο με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε έκτακτες περιπτώσεις. Αυτή είναι και η θέση του Κοινοβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια και περιλαμβάνεται στη γνωμοδότησή μας. Επίσης, προτείνουμε να συμπεριληφθεί μία αναφορά στην οποία θα ζητείτε μια εξαίρεση σε περίπτωση προγραμμάτων που εγκρίνονται εξαίρετα, όπως είναι το 2013. Κατά εξαίρεση, με συγχωρείτε. Ούτως ώστε να μην έχουμε ένα άνισο προφίλ και στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που δεν έχω κάνει είναι ότι δεν έχουμε τροποποιήσει τα κριτήρια για τα επιδόματα ή τη διανομή ανάμεσα στις διαφορετικές περιφέρειες και επίσης δεν έχουμε τροποποιήσει τους ε, γενικούς στόχους συνοχής όλων των τύπων ε, που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Συνοχής. Με τους υπόλοιπους συντενιστές, όπως σας είπα, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε ζητήματα προϋπολογισμού και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα εθνικά ζητήματα. Επομένως, ούτε πήραμε ούτε δώσαμε χρήματα. Δεν προτείνουμε δηλαδή να δοθούν περισσότερα χρήματα σε συγκεκριμένες χώρες. Σε γενικές γραμμές, αυτό που έκανα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ήταν να μεταφράσω σε νούμερα, σε ζητήματα προϋπολογισμού, αυτά τα οποία αποφασίσαμε τον Μάρτιο όπως συμφωνήσαμε από κοινού οι συντονιστές, αποφασίσαμε να διατηρηθεί το επίπεδο της ε, συγχρηματοδότησης, να αυξηθούν τα επιδόματα για γεωγραφική συνεργασία. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, πίστευω ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν έχει αντιφάσεις. Ε, μέχρι την 3η Νοεμβρίου μπορείτε να υποβάλλετε τις προτάσεις σας, ούτως ώστε να κατατεθεί την 5η Νοεμβρίου στην Επιτροπή. Περιμένω να υιοθετηθεί ομόφωνα, αλλά βεβαίω είμαι ανοιχτό σε οποιασδήποτε προτάσεις, σχόλια έχετε να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζικφρίτ. Δεν βλέπω. Υπάρχει εδώ. Έχουμε σκιώδη συγκητή από τους σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ, η Άιντα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι προφανώς και θα καταθέσουμε κάποιες ε, τροπολογίες, αλλά όπως είπε και ο συνδηγητής, ε, παρακολουθεί μόνος έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που έχουν σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ως εκ τούτου δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα όσο δεν είναι εδώ ε, παρόν ο κύριος Ουλμπριχτ, εκτός αν ο κύριος Φερνάντες ε, θέλει να λάβει το λόγο. Αν δεν θέλουμε να το λάβει το λόγο ο κύριος Φερνάντες, καλύτερα να πάμε πίσω στα κτίρια. Ε, αλλιώς θα πάμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Ολμπριχτ που έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής. Εγώ να σας πω και κάτι άλλο έτσι για να περνάει και η ώρα θα ήθελα να μιλήσουμε για το κτίριο GMO2. JMO2. Ε, και να σας πω ποια είναι η κατάσταση. Ως Επιτροπή Προπολογισμών είχαμε ζητήσει να ενημερωθούμε επακριβώς για την ε, αύξηση κόστους, για τις αλλαγές και το τι ακριβώς θα λάβει η χώρα. Έχουμε τώρα τη σχετική πρόταση, έχουμε και τα απαραίτητα έγγραφα και η UL έχει καταθέσει και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν θέλω βέβαια να αναφερθώ σε αυτές γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όμως όλοι σας μπορείτε να δείτε με κάθε λεπτομέρεια τι άλλαξε και πώς ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι τον Ιούλιο του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Ε, στην αρχή προβλεπόταν 23 Ιουλίου, ε, τώρα όμως ε, προβλέπεται τον Φεβρουάριο του 2023 και η δεύτερη φάση τον Φεβρουάριο του 2024. Δηλαδή θα έχουμε μία καθυστέρηση τεσσάρων ετών η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τους εργολάβους, έπρεπε να συνευτούν ε, πολλά νέα συμβόλαια και μετά υπήρξε μία συμφωνία ανάμεσα στην κυρία Γεωργίεβα και τον κύριο Ασελμπόρν. Και αυτό οδήγησε στο ότι παρετηθήκαμε από ένα κέντρο υπολογισμών. Αυτό θα εγκατασταθεί κάπου αλλού. Έπρεπε να προσαρμοστεί το σχέδιο 3.700 θα είναι τώρα οι συνεργάτες και όχι 3.040. Αυτοί οι 3.700 θα είναι όλοι στο ίδιο κτίριο. Αυτό βέβαια θα είναι πιο δαπανηρό αλλά και πιο αποτελεσματικό. Ε, βεβαίως αυτό το κέντρο των υπολογισμών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών επίσης ε, αυτό σας είπα ότι θα εγκατασταθεί σε, σε κάποιο άλλο χώρο και εμείς το δεχτήκαμε αυτό. Κατόπιν υπήρξαν οι επιθέσεις στις Βρυξέλλες. Που τι συνέμενε αυτό? Συνέμενε ότι θα έπρεπε να εξεταστούν όλα τα κτίρια κάτω από το πρίσμα της ασφάλειας. Άρα και αυτό. Έγινε λοιπόν μια μελέτη σκοπιμότητας. Ε, λήφθησαν υπόψη στον προγραμματισμό όλες οι απαραίτητες ε, διαστάσεις περί ασφάλειας, γιατί δεν έχει νόημα να μπαίνει κανείς σε ένα κτίριο και μετά από λίγο να πρέπει να μετακομίσει γιατί δεν είναι ασφαλές. 17,1 εκατομμύρια είναι το κόστος αποτελούνται από δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά τις, ε, τα θέματα ασφάλειας και το δεύτερο αφορά περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με την εγκατάσταση των ε, συνεργατών και την εξαίρεση του κέντρου υπολογιστών. Έχουμε όμως και μία εξοικονόμηση, λόγω ακριβώς του ότι θα εγκατασταθεί κάπου αλλού το κέντρο των υπολογιστών. Έχουμε ε, και ένα σχετικό απόθεμα, ε, το οποίο αρχικά ήταν το 10% του προγράμματος. 350 εκατομμύρια ευρώ ήταν το αρχικό, ε, αρχικός, αρχική πρόβλεψη 345 εκατομμύρια ήταν το ανώτατο όριο και αν δούμε λιγάκι τους υπολογισμούς συμπεριλαμβάνοντας και το κόστος ασφάλειας όπως ακριβώς το ανέφερα προηγουμένως νομίζω ότι από αυτού μπορούμε να συμφωνήσουμε αύριο γιατί σε τελική ανάλυση πάνω ε, θα εγκατσατούν στο κτίριο περισσότεροι άλλοι 600 ε, υπάλληλοι χωρίς όμως να προκληθεί ουσιαστικό κόστος ε, στο κτίριο. Άρα μιλάμε για αποτελεσματικότητα. Και ελπίζω πλέον το κτίριο αυτό να είναι έτοιμο το 2024 και μην να, μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Εύχομαι καλή τύχη. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θέλουν να πούν κάτι. Από ό,τι βλέπω όχι. Ε, βλέπω ότι ήρθε και ο συνάδελφος κύριος Ουλμπριχτ. Γιάν. Είσαι ο εισηγητής ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής και σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δουλεύουμε παράλληλα για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και για τα ε, για, τις, ε, λεγό, για τους λεγόμενους τομεακούς ε, κανονισμούς μεταξύ των οποίων και αυτό της Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής μαζί με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το σημαντικό είναι αυτό το σχέδιο το οποίο υπέβαλε η Κομισιόν είναι ότι προσπαθεί να αλλάξει η Κομισιόν την στρατηγική της με τρόπον ώστε να Διαβρύνουν το πεδίο εφαρμογής ε, των παρεμβάσεων του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όχι μόνο για τις λιγότερο αναπτυγμένες, αλλά και για τις περισσότερο αναπτυγμένες ε, περιφέρειες. Αυτό είναι το πρώτο που θέλουν να κάνουν. Θέλουν λοιπόν να αλλάξουν και τις στατιστικές. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, ε, διότι υπάρχουν δύο ειδών στατιστικές που προτείνονται. Στατιστικές οι οποίες βασίζονται στο ΑΕΠ, ε, κατά σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2, το λεγόμενο περιφερειακό δηλαδή, και ε, αυτή η στατιστική βρίσκεται και στην, ε, στον κανονισμό CPR, αλλά έχουμε όμως και μία άλλη πρόταση, η οποία θα είναι η εξής. Θα βασίζεται στο εθνικό εισόδημα, σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό το επίπεδο εθνικού εισοδήματος θα χρησιμοποιηθεί σε ε, όρους θεματικής ε, ε, αναφοράς. Μέχρι τώρα όμως αυτό βασιζόταν στον ΝΑΤΣ 2 ΑΕΠ κατά κεφαλή, ενώ τώρα αλλάζει και γίνεται πρόταση όπως και στο Ταμείο Συνοχής να γίνεται ο υπολογισμός βάσει το εθνικό εισόδημα και αναπεριφέρεια. Η Κομισιόν πρότεινε να χρησιμοποιήσει ε, τον ίδιο τρόπο για τις λιγότερο αναπτυγμένες, περισσότερο αναπτυγμένες και σε μετάβαση. Ε, και ε, επομένως όλα αυτά γίνονται ιδιαίτερα περίπλοκα γιατί κανείς δεν καταλαβαίνει πλέον περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω το εξής, να χρησιμοποιηθεί η θεματική συγκέντρωση μονάχα σε δύο επίπεδα ε, βασιζόμενα δηλαδή το εθνικό εισόδημα, έτσι όπως αυτό χρησιμοποιείται για το Ταμείο Συνοχής. Προτείνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε μία κατηγορία για τις χώρες συνοχής και μία κατηγορία για τις χώρες μη συνοχής, τελεία και παύλα, έτσι ώστε τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Η θεματική συγκέντρωση σε αυτό το επίπεδο να γίνεται λοιπόν με βάση του εθνικού εισοδήματος και όχι του ΑΕΠ. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να έχουμε δύο ομάδες, ε, ε, ένα και δύο αλλά έχουμε και μια δεύτερη πρόταση ε, να προχωρήσουμε βάσει των λεγόμενων POs, δηλαδή των στόχων προτεραιότητας. Στην πρόταση τη νέα της Κομισιόν έχουμε δύο νέους τέτοιους POs, ε, στόχους προτεραιότητας και αυτό είναι αμφιλεγόμενο γιατί ε, ο πρώτος PO α πούμε αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση, με την καινοτομία κλπ. Ο δεύτερος αφορά την κλιματική αλλαγή. Ο τρίτος στόχος προτεραιότητας αφορά την ε, κινητικότητα και την ε, διασύνδεση και διασυνδεσιμότητα, εν πάση Ε, υπάρχουν και κάποιες άλλες POs ε, που αφορούν όμως τοπικές δράσεις. Εγώ προτείνω να χρησιμοποιήσουμε τη θεματική συγκέντρωση βασιζόμενη στους δύο πρώτους ε, στόχους POs, ε, δηλαδή καινοτομία και ψηφιοποίηση και έρευνα. Στα πλαίσια της ε, πολιτικής σύνοχης και, στο, και να χρησιμοποιήσουμε και τον δεύτερο στόχο, στο δεύτερο στοιχείο που αφορά την κλιματική αλλαγή. Το αμφιλεγόμενο είναι ότι η ψηφιοποίηση δεν περιλαμβάνεται ε, στις ε, ε, οι προτεραιότητες διότι συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο ενέχεται στην διασυνδεσιμότητα. Εγώ προτείνω λοιπόν την ψηφιοποίηση να τη βάλουμε στο, στο πρώτο στοιχείο και αν πραγματικά θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό τότε και η ψηφιοποίηση θα πρέπει να περθεί στο πρώτο στοιχείο. Επίσης η κινητικότητα είναι κάτι σημαντικό αλλά η κινητικότητα δεν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες στις δύο πρώτες προτεραιότητες ε, και η κλιματική αλλαγή είναι στο 2. Προτείνω λοιπόν να αλλάξουμε τη θέση της κινητικότητας και να τη βάλουμε στο 2. Δηλαδή να προτείνουμε πρώτον να αλλάξουμε τα κριτήρια για τη θεματική συγκέντρωση χρησιμοποιώντα μονάχα δύο ε, ομάδε, χώρε συνοχή από τη μία, μη συνοχή από την άλλη. Και δεύτερον, να μεταφέρουμε την, την αστική κινητικότητα πιο πάνω και μια τρίτη πρόταση είναι να δούμε τα κριτήρια, τι είδους συγκέντρωση θέλουμε. Η Κομισιόν αυτό που προτείνει τώρα είναι το εξή. Οι πιο αναπτυγμένε χώρες, οι πιο αναπτυγμένε χώρες τονίζω, να έχουν 85% ε, ε, συγκέντρωση, δηλαδή μικρή ευελιξία. Εγώ προτείνω για τις χώρες μη συνοχής ε, να είναι 50% και για τις χώρες συνοχής να είναι 30% και νομίζω ότι για να, το καταλάβουν και οι συνάδελφοι θα σας δώσω το παράδειγμα της Φιλανδίας. Η Φιλανδία αυτή τη στιγμή, σήμερα, λόγω του ότι τα κριτήρια ε, το κριτήριο για τις ε, χώρες, ε, ε, για τις χώρες σε μετάβαση είναι το ΝΑΤΣ 2 ΑΕΠ, είναι στην ομάδα 2. Αλλά η Φιλανδία για την άλλη περίπτωση, σαν χώρα δηλαδή, είναι στις αναπτυγμένες. Επομένως έχουμε τις περιφέρειες οι οποίες είναι σε μετάβαση, ενώ τη χώρα η οποία είναι στις αναπτυγμένες χώρες. Smallest. Η ευελιξία θα πρέπει να αφορά τις μικρότερες ε, ε, χώρες ε, γιατί καταλαβαίνετε, γι' αυτό είπα και από την αρχή ότι οι στατιστικές είναι πολύ σημαντικές. Οι στατιστικές έτσι όπως χρησιμοποιούνται αλλοιώνουν την εικόνα. Γαλλία, άλλο παράδειγμα. Οι περισσότερες περιφέρειες στη Γαλλία θα είναι περιοχές σε μετάβαση. Αλλά εάν μιλήσουμε με όρους εισοδήματος τότε αλλάζει η κατάσταση. Μπερδεύεται λοιπόν η εικόνα. Επομένως επαναλαμβάνω για να καταλάβετε. Απλοποίηση πρώτα, απλούστευση, δύο ομάδες μόνο, μία, χώρα, μία ομάδα οι ε, χώρες συνοχής με ε, συγκέντρωση 30% και μη συνοχής με συγκέντρωση 50%. Επίσης, να βάλουμε και την ψηφιοποίηση ε, στον πρώτο ποιόου και στο δεύτερο ποιόου να βάλουμε εκτός από την κλιματική αλλαγή και την πρόθεση της πολυτροπικής, αστικής ε, και περιαστικής κινητικότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις ε, καλές ε, τις καλές εμπειρίες που έχουμε με τα λεγόμενα σε αυτές τις συμπράξεις. Λειτουργούν πάρα πολύ καλά στα πλαίσια του Τομείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της καταχώρησης των πόρων του και θεωρούμε ότι και η περιοχή, η Επιτροπή Περιφερειών αλλά και η ΕΟΚΕ ε, συμφωνούν με αυτό και εγώ προτείνω να πάμε στο 10% από το 5% στο 10%. Δεν θα σημάνει περισσότερα χρήματα, απλώς ε, ε, περί, ε, ε, απλώς ε, τα χρήματα τα οποία, τα κονδύλια τα οποία δίνονται αφορούν πιο συγκεκριμένες καταστάσεις. Περιγράφονται δηλαδή καλύτερα προγράμματα όχι στην τάξη του 5% του Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης αλλά στο 10%. Αυτά προτείνω λοιπόν στην γνωμοδότησή μα, η οποία θα πάει στην Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη ε, ω γνωμοδότηση τη δική μα Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, και ο ε, η Άιντα να λαμβάνει. Σε ευχαριστούμε Άιντα για αυτό που μα προσφέρει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι. Ε, τι να κάνω. Σήμερα η μοίρα το έχει να είμαι συνέχεια Εκπρόσωπο, τη ομάδα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τις προτάσει του κ. Όλμπρεχτ και χωρί ε, να είμαι ιδιαίτερα εμπειρογνώμων περί τα θέματα αυτά, νομίζω ότι προτείνει πολύ λογικά πράγματα. Ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό και αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να λάβει χώρα στην ε, ΡΕΤΖΙ, η οποία είναι και αρμόδια ε, απλούστευση των κατηγοριών, ε, μετατόπιση θεμάτων εντός των κατηγοριών, ε, νομίζω ότι ε, ο ίδιος ξέρει πάρα πολύ καλά και την πολιτική συνοχή και επομένως ε, θεωρώ ότι πολύ καλά τα λέει, δεν έχω κανένα λόγο να αντιδράσω, αλλά γιατί να συζητιέται το θέμα αυτό εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Άιντα. Από τις άλλες πολιτικές ομάδες, από το ECR, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ούλμπριχ. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να εξορθολογήσουμε διαδικασίες, να δημιουργήσουμε κατηγορίες, γιατί με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η διαφάνεια. Επανειλημμένα, αντιμετωπίζουμε αιτιάσεις ότι οι πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Και αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι τα θέματα είναι περίπλοκα, το κάνουμε και πείτε λιγάκι αυτό, αλλά στη τελική ανάλυση όλοι λέμε ότι ο στόχος μας είναι να υπάρχει διαφάνεια. Εγώ θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και το στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Γιάν, θέλει εσύ το λόγο? Το ζήτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε ως Επιτροπή Προεπολογισμού. Δεν είναι μια τμηματική απόφαση. Η συζήτησή μας έχει να κάνει με τον προπολογισμό. Τι έχουμε να πούμε όμως πάνω στον προπολογισμό και πολλά, γιατί δεν συζητάμε ε, πόσα χρήματα προτείνει για το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη η Επιτροπή Περιφερειών. Δεν συζητάμε τις προτάσεις τη ε, Ρέτζη, αν μιλάμε για περισσότερα ή λιγότερα χρήματα. Πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα, ε, σε αυτό μπορούμε να κάνουμε ότι δηλαδή τα κριτήρια των της χρήσης των ε, Ευρωπαϊκών Ταμείων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, γιατί αυτό είναι ζήτημα απλότητας, διαφάνειας κτλ. Αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν είναι ότι αν έλθουμε σε λεπτομέρειε οι καταστάσεις δεν είναι ίδιε, αλλά όταν κοιτάζουμε τι στατιστικέ και πώ διανέμουμε τα χρήματα, ο τρόπο που διανέμουμε τα χρήματα, αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, αυτό θα πρέπει να είναι απλό, προφανέ. Γι' αυτό το λόγο, στην περίπτωση αυτή, η γνωμοδότηση έγκυται σε εμά, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θέλω να σας υπενθυμίσω, Πρόεδρε, ότι υπάρχει συμφωνία, η συμφωνία της συνεδρίασης των Πρόεδρων. Σύμφωνα με τη συμφωνία αυτήν, κανένας από τους κανονισμούς δεν μπορεί να ψηφιστεί στις επιτροπές προτού ψηφιστεί στην Ολομέλεια το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ισχύει και για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για το Ταμείο Συνοχής. Τα χρήματα αυτά θα βρίσκονται μέσα στον κανονισμό. Γι' αυτό το λόγο δεν ε, μπορώ να, να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα στην ονομοδότηση. Γιατί θεωρώ ότι θα είναι απόφαση του ψηφίσματος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σας ευχαριστώ. Και εμεί ευχαριστούμε πολύ Γιάν. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να λάβει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εισηγητή και τους συναδέλφους. Και θα ήθελα τώρα να επανέλθουμε ε, στην κτηριακή πολιτική, αγαπητέ Ζεράρ Ντεπρέ. ενημερώσαμε ήδη για τρία κτίρια. Έχουμε συζητήσει τρεις κτηριακές εκθέσεις. Παρακαλώ, Γιάννη. επειδή η γνωμοδότησή μας είναι ένα νομοθετικό κτίριο, ε, κείμενο, με συγχωρείτε, μπορεί να, να επιστρέφουν τροπολογίες. Υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικό για το Ταμείο Συνοχής που έχει να κάνει με τη μείωση του αποθέματος. Αυτό είναι μια αλλαγή στην πολιτική. Κάτι το οποίο συζητάμε στην Επιτροπή Προπολογισμού, συζητάμε στην Επιτροπή των Περιφορίων, ρωτάμε τι έγινε, γιατί μειώθηκε κατά 46% το Ταμείο της Συνοχής και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Διότι για πολιτικούς λόγους είχε φουσκωθεί το ποσό αυτό, φαινόταν παραπάνω. Είχαμε λοιπόν κάτι το οποίο ήταν τεχνητά υψηλότερο. Τώρα θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότατα. Είναι σημαντική και αυτή η πληροφορία, θεωρώ εγώ. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τη μείωση του 46% για να επιστρέψουμε σε κανονικά επίπεδα σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής. Δεν είναι ένα νομοθετικό κείμενο. Θα περιλαμβάνεται όμως στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας ε, είπατε. Δεν ξέρω, ε, θέλετε να παρατηρήσετε κάτι, θέλετε να προσθέσετε, υπάρχει κάτι άλλο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για κατάθεση, η καταληκτική προθεσμία, η κατάθεση τροπολογιών είναι τον Οκτώβρη, 1η Οκτωβρίου στις 3 ε, ώρα το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε στις 5 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Αγαπητέ Ζεράρ, ε, και προηγουμένως απευθύνθηκα σε σένα. Σήμερα δεν έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Επιτροπή μας και έχουμε ήδη συζητήσει για τρία κτίρια. Τώρα, εσύ είσαι σκιώδης συγητής. Αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι, μπορεί να το κάνεις. Ασχοληθήκαμε το Πασός και εσύ είχες ε, κάνει το ερώτημα ε, πώς ακριβώς θα χρησιμοποιείτε το Πασός. Τι είδου συνεδριάσει ε, θα φιλοξενεί το κτίριο αυτό. Το Κοινοβούλιο έχει απαντήσει. Αν θέλει όμω να ξανακούσει την απάντηση, ευχαρίστω να την επαναλάβουμε. Κυρία Πρόεδρε, όχι όσον αφορά το κτίριο Μπαζός. Δεν έχω αντίρρηση. Ε, σε σχέση με αυτά που γίνονται και οργανώνονται στο Ζαμονέ ε, ε, και το, μάλλον τον οίκο Ζαμονέ απλώς το μπαζός τελικά είναι ακριβό Νομίζω ότι παρότι είναι πιο ακριβά, ξέρω τα οι τιμές οι πιο ακριβές στο Λουξεμβούργο, εδώ είναι πολύ ακριβά ανά τετραγωνικό μέτρο. Ε, και εν πάση περιπτώσει, ναι, τι, αν θέλει κάποιο να επενδύσει, δηλαδή να αγοράσει ε, οικόπεδο στον σου. Αγαπητέ Ζεράρ, θέλω να πω, 1200 ε, τετραγωνικά για 260.000 ευρώ ούτε στις Βρυξέλλες δεν μπορεί κανείς να τα βρει. Για να μην πούμε τώρα Μόναχο, Παρίσι, Λονδίνο, Ξέχνατε αυτά. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Πολύ ωραία. Ε, Έχουμε τώρα το κτίριο Eurofis ε, στο Λουξεμβούργο. Συζητήσαμε και γι' αυτό. Αν δεν έχεις κάποια ερώτηση επ' αυτού. Και επίσης ε, συζητήσαμε και για το κτίριο GMO2 στο Λουξεμβούργο. Ε, και θα ήθελα τώρα να περάσω στο ΕΣΜΑ. Αυτή τη στιγμή η ΕΣΜΑ βρίσκεται στην Κρενέλ, πρώτο, τρίτος και τέταρτος όροφο στο Παρίσι. Δύο φορές ε, είχαμε επέκταση ε, λόγω του ότι αυξήθηκαν ε, οι δαπάνες. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. 275 είναι οι εργαζόμενοι στο κτίριο αυτό, οι οποίοι εργάζονται σε 6.400 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Τα 4.500 είναι για εσωτερική χρήση και τα 1.500 που υπολείπονται προσφέρονται στο κτίριο για εξωτερική χρήση. Υπάρχει και κάποια έκθεση όπου είναι εγκατεστημένα τα αρχεία. Ανάτομο 23 τετραγωνικά, το ετήσιο κόστος 5,160 εκατομμύρια ευρώ και αυτό σημαίνει ανά τετραγωνικό 795,72 ευρώ. Το Παρίσι πάντα ήταν πιο προσιτό, ηρωνικά βέβαια το λέω, το Παρίσι και το Λονδίνο ε, βεβαίως πάντα μας δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τα μισθώματα. Χρειαζόμαστε νέο κτίριο για το κτίριο ΕΑΚΑ ε, και γι' αυτό θέλουμε να ενοικιάσουμε το κτίριο iBox ε, στο Παρίσι, ε, κάποιους ορόφους αυτού του κτιρίου. Το κτίριο αυτό αυτή τη στιγμή είναι υπό ανακαίνιση, προέρχεται από το 1900 74 ε, τότε πρωτοσυνήφθη το πρώτο συμβόλαιο. Ε, το 2019 θα υπάρξουν κάποιες παρατάσεις του Συμβουλίου αν το επιθυμούμε. Υπάρχει μία ρήτρα όπου ε, αν υπάρξει κάποια καθυστέρηση ο ιδιοκτήτης βέβαια λέει ότι δεν θα υπάρξει καμιά σημαντική καθυστέρηση και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά που έχουμε ανακαινήσεις έχουμε και καθυστερήσεις. το κτίριο αυτό, μάλλον η ΕΚΑ έχει διαπραγματευτεί ρήτρα καταγγελίας έξι χρόνια ε, και σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το μίστομα και εκεί προβλέπονται σχετικές ρυθμίσεις. Ε, προβλέπεται βέβαια και το ότι αν υπάρξει κάποια επέκταση και το ζητήσει ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση 4, τόσα εκατομμύρια. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό, αλλά πάντα πρέπει να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Συνολική έκταση 9.200 τετραγωνικά μέτρα ε, σε 17 περίπου ορόφους. 8.000 τόσα τετραγωνικά μέτρα είναι αυτά που έχουμε νοικιάσει και όπως σας είπα ένα μεγάλο κομμάτι εξ αυτών χρησιμοποιούνται για κτίρια, για meeting, η ΕΣΜΑ χρειάζεται ε, πάρα πολλές αίθουσες ε, για meetings και συνεδριάσεις γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις με ασφάλειες ε, των οποίων προείσταται, ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλα. Υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Ε, το 2022 ε, θα εγκατασταθούν στο κτίριο 703 υπάλληλοι, 703 πάρα πολύ, δεν είναι. 250 ήταν τόσοι μέχρι τώρα. 700, τώρα πώς πάμε από τους 250 στους 700. Μήπως είναι τυπογραφικό το λάθος. Ε, με βάση της ε, νέας προτινόμενης ε, νομοθεσίας ίσως γύρω στους 450 να είναι οι υπάλληλοι, το πολύ, 450. Μάλλον δηλαδή τυπογραφικό το λάθος. Το ετήσιο μίστομα 4,933 εκατομμύρια προβλέπονται κάποιες απαλλαγές και Πέντε ε, μηνιαία μισθώματα. Ε, έχουμε κάποια εξοικονόμηση αν αυτά καταβληθούν ε, προκαταβολικά. Έχουμε εργασίες ανακαίνησης 5,4 εκατομμύρια. Αυτά βέβαια τα αναλαμβάνει ο εκμισθωτής. Ως εκ τούτου μειώνεται το κόστος του μισθώματος και το ετήσιο ε, συνολικό κόστος, αν τα συνυπολογίσει όλα, πάγιες δαπάνες και όλα τα υπόλοιπα, 5,927 εκατομμύρια. Με βάση το ότι θα έχουμε αύξηση προσωπικού ε, στον ίδιο χώρο και σε σύγκριση με το προηγούμενο κτίριο, που βέβαια δεν μας ικανοποιεί πλέον, έχουμε μία αύξηση της τάξης των 800.000. Λογικό μου φαίνεται αυτό γιατί θα εγκαταστήσουμε περισσότερο προσωπικό σε ανακαινισμένο κτίριο. Εδώ περιλαμβάνεται και το κόστος ανακαίνησης. Νομίζω ότι η ΕΣΜΑ τα έκανε πάρα πολύ καλά. Από 43 αρχικές προσφορές επέλεξε 22 που κάλυπταν τα κριτήριά της. Είχε και επαφές με τη γαλλική κυβέρνηση. Αυτή βέβαια δεν μπορούσε να διαθέσει κτίρια. Ως εκ τούτου η ΕΣΜΑ πραγματικά ασχολήθηκε ουσιαστικά με την κτηριακή πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό για το Παρίσι είναι η βέλτιστη δυνατή λύση. Εκ μέρους των σοσιαλδημοκρατών δεν ξέρω αν έχει κανείς να παρατηρήσει κάτι. Από ό,τι βλέπω όχι. Ζεράρ, εσύ θέλεις να μιλήσεις εκ μέρους των φιλελευθέρων. Όχι, δεν θα, δεν θα μιλήσω σε πρόσωπο τη ΑΛΔΕ, αλλά ε, ως, ε, θα κάνω προσωπικές παρατήρησει. Ε, ε, υπάρχουν επιπλέον τετραγωνικά προ και βλέπω ότι θα υπάρχουν εκεί περισσότερες θέσεις πάρκινγκ για τα ποδήλατα παρά για τα αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό και έπρεπε να το σημειώσω οπωσδήποτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω κάτι, για δοκιμάστε, εγώ το λέω σε όλους. Πηγαίνετε με το αυτοκίνητο στο Παρίσι. Αν δεν έχει συνηθίσει κανείς να οδηγεί αυτοκίνητο στο Παρίσι, η εμπειρία είναι τραυματική. Ακριβώς όπως και στη Ρώμη. Αλλά, ωραία, σωστά το επισήμανες. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις προς την ΕΣΜΑ. Αύριο θα ψηφίσουμε. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή δουλειά. Πάμε. Προκατρακτική ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προκατακτική ενημέρωση αντιπροσωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Πακού στο Αζερμπαϊτζάν. 1.200 τόσα τετραγωνικά μέτρα στον 11ο όροφο ενό κτηρίου 22 ορόφων. Αυτό θα νοικιάσουμε. Το ετήσιο κόστος ε, θα είναι 828.000 ευρώ. Έχουμε μία προσφορά, μακροχρόνια μίσθωση ε, αυτό το ε, προσφέρει ο Αυτή τη στιγμή γίνεται ενδελεχής εξέταση του ε, συμβολέου. Ε, το κτίριο βρίσκεται στην στη δυνατή θέση, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και προσφέρει τη δυνατότητα υπενικίασης. Ως εκ τούτου φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Και υπάρχει και μία προκατακτική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κτίριο Λουά 78 και Λουά 82. Όσον αφορά το Λουά 78, εδώ έχουμε ε, ένα συγκρότημα που αποτελείται από 8 κατ' ε, ε, κτίρια, εκ των οποίων τα έξι βρίσκονται ήδη στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται τα κτίρια της από το 2025 να τα ε, ανακαινήσει σε δύο φάσεις, γιατί πολλά κτίρια έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους και χρειάζονται ανακαίνιση εκβάθρων. Ε, το ΛΟΑ ε, 86 ε, έχουμε και άλλα κτίρια, το 100 και πάρα πολλά άλλα. Αυτά προβλέπεται όλα να ανακαινιστούν μέχρι το 2025 κατά τη δεύτερη φάση ε, το κτίριο ΛΟΑ 79 ε, το 78 και το 88 αυτά θα ανακαινιστούν μέχρι το έτος 2030. Και όλα αυτά θα γίνουν σε συνεργασία με την πόλη των Βρυξελών και την κυβέρνηση. Τον Μάρτιο του 2018 Είχαμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τα κτίρια ε, ΛΟΑ 130 και εκεί ε, προβλέπθηκε εκτός από την ανακαίνιση να προσθεθούν και άλλα δύο κτίρια για να υπάρχει καλύτερη ένταξη στην εικόνα της πόλης. Αυτός είναι ο στόχος ε, όσον αφορά το ΛΟΑ 80, το 82 μάλλον, εκεί μιλάμε και για χώρους άθμευσης στο υπόγειο. Αυτή τη στιγμή ε, τα συμβόλαια ε, προβλέπονται μέχρι το 2027 και κατόπιν εκπνέουν. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς ε, να ρωτήσει κάτι εκ μέρους των σοσιαλδημοκρατών, των φιλελευθέρων, του ECR. Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν έχει να ρωτήσει τίποτα και αύριο στις 4 η ώρα θα ψηφίσουμε για την κτηριακή πολιτική, ε, για όλα τα κτίρια. Και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους σοσιαλδημοκράτες, ε, παρακαλώ να μας θέσετε τα ερωτήματα αυτά ή αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με όσους ήταν ε, σήμερα εδώ στη συνεδρίαση για να σας ενημερώσουν. Πολύ ωραία. Αύριο το πρωί έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικής και Αναπτυματικής Πολιτικής στις 10.30. Είναι το, η ακρόαση για το ΕΨΙ και μετά έχουμε και άλλη ακρόαση στις 2.30. Ε, οι συντονιστές ε, θα συναντηθούν στις 5 ε, η ώρα, όχι στις 4.30. 4.30 θα συναντηθούν οι αρμόδιοι για ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποια άλλη ερώτηση από αυτού. Από ό,τι βλέπω, όχι. Ως εκ τούτου, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ωραία.